Παρακαλώ λίγη ησυχία. Συνεχίζουμε με την ημερήσια διάταξη. Σημείο 7. Παρακαλώ, Σιλάνς. Τροποποίηση του κανονισμού 1198 του Συμβουλίου σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τις θαλάσσιες υποθέσεις και την αλία. Θα γίνει η παρουσίαση από τον εισηγητή μας, τον κύριο Καντέκ του εγγράφου εργασία που εκπώνησε και χωρί άλλη καθυστέρηση να δώσω το λόγο στον κύριο Καντέκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, το ΕΤΘΑ αποτελεί το οικονομικό σκέλο τη μεταρρύθμιση τη ΚΑΠ, αφορά και την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει 6 δισεκατομμύρια 500 εκατομμύρια για την περίοδο 2013-2020 και 342 εκατομμύρια για την ολοκληρωμένη θαλάσσια περιοχή, ε, πολιτική χωρίς το εξωτερικό σκέλος της ΚΑΠ και τις ε, οργανώσεις, περιφερειακές οργανώσεις που θα χρηματοδοτηθούν από άλλα ε, κονδύλια του προϋπολογισμού. Το χρονοδιάγραμμα που σας προτείνω λαμβάνει υπόψη την ανάγκη προηγούμενη συμφωνία για του δύο γενικού κανονισμού, κατά κάποιο τρόπο, από του οποίου εξαρτάται το ΕΤΘΑ, δηλαδή το βασικό κανονισμό της κοινή ελευθερική πολιτική και το Γενικό Κανονισμό για τα Διαρθρωτικά Ταμεία Αφετέρου. Ο δεύτερος αυτό κανονισμός εξετάζεται αυτή τη στιγμή στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Η υιοθέτηση του κανονισμού για το ΕΤΘΑ στην Επιτροπή Αλλία προβλέπεται να γίνει τον Νοέμβριο του 2012, ενώ η ψηφοφορία στην Ολομέλεια θα γίνει τον Ιανουάριο του 2013. Είπαμε επανειλημμένως ότι διαφωνώ με κάποιες προτάσεις της μεταρρύθμισης ελευτικής πολιτικής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οπότε είναι λογικό κάποιε προτάσει μου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θαλάσσιων Υποθέσεων και Αλία να μην ευθυγραμμίζονται με τι προτάσει Ευρωπαϊκή Επιτροπής στο βασικό κανονισμό. Όλοι γνωρίζουν ότι είμαι υπέρ μεγάλη μεταρρύθμιση του βασικού κανονισμού, γιατί αλλιώ το ΕΤΘΑ ουσιαστικά θα βοηθήσει στην πάυση της αλληλευτική ε, δραστηριότητας, σε μια ανεπιθύμητη επέμβαση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δικαιολογεί την πρόταση μεταρρύθμισης ε, βεβαιώνοντας ότι θα περιορίσει την πλεονάζουσα αλληλευτική ικανότητα με στόχο να περιοριστεί ο αλληλευτικό στόλο, είναι αμφισβητήσιμο όμω ο χαρακτήρα αυτή τη διατύπωση. Η πλεονάζουσα αλληλευτική ικανότητα δεν έχει προσδιοριστεί από την Επιτροπή μέχρι σήμερα. Επομένω, είναι δύσκολο να αποδειχθεί μια τέτοια πλεονάζουσα αλληλευτική ικανότητα. Ακόμη και αν είναι πιθανό ορισμένε περιοχέ να διαθέτουν πολύ αυξημένη αλληλευτική ικανότητα ω προ του διαθέσιμου πόρου, αυτή η κατάσταση δεν πάβει να είναι αποσπασματική και χωρικά περιορισμένη και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να επεκταθεί σε όλε τι ελευτικέ περιοχέ Ένωση, ούτε να εκλειφθεί ω αξίωμα. Μάλιστα σήμερα το πρωί υπενθύμησε ότι θα πρέπει να συγχαίουμε την αλληλευτική ε, ικανότητα ε, που αποτιμάται σε κιλοβατόρες και την αλληλευτική προσπάθεια που αποτιμάται σε τόνους αλλιεύματος. Ε, άλλο πλεονάζω αλληλευτική ικανότητα και άλλο υπεραλίευση. Σε μερικές περιπτώσεις συμπίπτουν βέβαια, αλλά δεν ταυτίζονται. Θα ήθελα πάντως να μην στηρίξουμε μία μεταρρύθμιση πάνω σε μία απλή διαβεβαίωση που στερείται συγκεκριμένη νομική ή επιστημονική βάση. Είναι απαραίτητο να εξολογιστεί συγκεκριμένα η αλληλευτική αξιολογηθει συγκεκριμενα η ελευτικη ικανοτητα του ευρωπαϊκού στόλου, Προτελουθούν πιθανέ ενέργειε για αυτόν τον παράγοντα. Εξάλλου αυτή η βούληση να μειωθεί η υποτιθέμενη πλεονάσου αλλιευτική ικανότητα του στόλου δεν θα έχει καμία επίδραση σε αλλιευμένε ποσότητε. Σε αντίθεση με όσα είχε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο βαθμό που αυτέ εξακολουθούσαν εξαρτώνται από τα συνολικά επιτρεπόμενα αλλιεύματα, τα ΤΑΚ και τι καθορισμένε αιτήσει ποσοστώσει. Διαπιστώνω λοιπόν ότι η Επιτροπή προτείνει να αλλιεύεται η ίδια ποσότητα ηχθείων από μικρότερο αριθμό αλλιευτικών σκαφών, θέτοντα έτσι σε κίνδυνο πολύ άριθμε αλλιευτικέ επιχειρήσει, ιδίω μικρή κλίμακα ή και συνεπώ πολλέ θέσει εργασία. Όπω γνωρίζετε, αφισβητώ αυτή την κατεύθυνση. Το κυρίαρχο μέτρο που προτείνεται στο βασικό κανονισμό για να περιοριστεί η υποτιθέμενη σε αλληλευτική ικανότητα είναι η θέσπιση μεταβιβάσιμων αδειών αλεία ή αλληλευτικών παραχωρήσεων. Η αναπόφευκτη συνέπεια αυτή τη διάταξη θα ήταν η συγκέντρωση αλληλευτικών δικαιωμάτων στα χέρια ενό μικρού αριθμού επιχειρηματιών. Αυτή η διάταξη θα έθετε σε κίνδυνο τη μικρή κλίμακα αλεία αφήνοντα ελεύθερο το πεδίο μόνο στι αγορέ που ξέρουμε που μα οδήγησαν σε άλλου τομεί. Η λογική συνέπεια τη καθιέρωση μεταβιβάσεων αλληλευτικών αδειών θα ήταν ένα προσανατολισμό του ΕΤΘΑ προ την ανασυγκρότηση των αλλιών εκτό του αλληλευτικού τομέα. Πράγμα το οποίο αποτυπώνεται ξεκάθαρα στο άρθρο 32. Αυτή η πρόταση θεσμοθετεί το προαναγγελθέν τέλο τη μικρή κλίμακα υπαράκτεια αλληλεία και επομένω ε, είναι απαράδεκτη, όπω ε, δήλωσαν και πολλοί ευρωβουλευτέ. Ο εισηγητή θεωρεί ότι αυτή η αλληλεία έχει μέρο στην Ευρώπη, ενώ μάλιστα η Ευρωπαϊκή Ένωση παράγει μόλι το 30% των προϊόντων αλληλεία και υδατοκαλλιέργεια που καταναλώνει και παραμένει ο πιο δεσμευτικό θαλάσσιο χώρο και η μεγαλύτερη αγορά του κόσμου. Ε, και ο πιο δεσμευτικό θαλάσσιο χώρο από άποψη προστασία των πόρων. Ένα φιλόδοξο ΕΤΘΑ είναι ασυμβίβαστο με την πρόταση βασικού κανονισμού όπω έχει υποβληθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από άποψη διαχείριση, προτείνω μια κοινή ελευτική πολιτική διαρθρωμένη πάνω σε τρία εργαλεία. Τη διατήρηση τη αρχή τη σχετική σταθερότητα, μέτρα περιορισμού των αλλιευμάτων και τη ελευτική προσπάθεια, τάκ δηλαδή και ποσοστό που προσδιορίζουν κάθε χρόνο τι αλλιευμένε ποσότητε, τεχνικά μέτρα που ρυθμίζουν τον αλλιευτικό εξοπλισμό για μεγαλύτερη επιλεκτικότητα. Αυτά τα τρία εργαλεία που συμπληρώνονται από καλύτερου ελέγχου και από διαρθρωτικέ ενέργειε στα πλαίσια του ΕΤΘΑ αποτελούν αποτελεσματικά εργαλεία για την διασφάλιση μια αηφόρου αλλιέ που θα επιτρέπει τη διαφύλαξη των πόρων, την προγραμματισμένη επίτευξη τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση και διατήρηση των εμπλεκόμενων δραστηριοτήτων και των θέσεων εργασία. Και έρχομαι τώρα στι προτάσει μου για το ΕΤΘΑ. Μία ενίσχυση του ελέγχου είναι απαραίτητη για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με του κανόνε τη κοινή αλληλευτική πολιτική και άρα η βιωσιμότητα τη αλληλεία. Χαίρομαι για τι προτάσει Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο άρθρο 78 που προβλέπει στήριξη των ελεκτικών προσπαθειών. Θα πρέπει επίσης να ενισχυθούν οι επιστημονικές πληροφορίες ό,τι αφορά την αποσωτική και ποιοτική κατάσταση των εκθιαποθεμάτων, ώστε να έχουμε ε, ποιοτικά επιστημονικά πορίσματα για όλα τα εκθιαποθέματα της Ένωσης. Και χαίρομαι για την θέση που δίνεται στην εταιρική σχέση επιστημόνων και αλλιέων σε ό,τι αφορά τη συγκέντρωση δεδομένων, μελετών και χρήση βέλτιστων πρακτικών και γνώσεων για να επιτύχουμε τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση το συντομότερο δυνατό για όλα τα εμπορικά είδη. Η συγκέντρωση δεδομένων αποτελεί, ε, έχει θεμελιώδη ρόλο. Προτείνω λοιπόν να ανέρθει στο 75% το ποσοστό χρηματοδότηση ε, στο άρθρο 79. Όπω ξέρετε, ο Ευρωπαϊκό Στόλο είναι γεράσκον. Το μέσο όρο τη ηλικία των πλοίων είναι 25 χρόνια, κάτι που δημιουργεί προβλήματα ασφάλεια στο κατάστρωμα και προβλήματα κατανάλωσης ε, καυσίμων. Θα θέλαμε με το ΕΤΘΑ να ενισχυθεί ο εξυγχρονισμός του στόλου υπό αυστηρές συνθήκες, ώστε να εθαρρύνουμε την καλύτερη αλίευση και όχι την ε, μεγαλύτερη αλίευση. Επίσης, να χρηματοδοτηθούν επενδύσεις για τον εξυγχρονισμό πλοίων και πάλι υπό για να βελτιωθούν οι εργασιακέ συνθήκε, η ασφάλεια, να περιοριστεί η κατανάλωση σε καύσιμα, η παραγωγή και να χρησιμοποιηθούν πιο επιλεκτικά αλληλευτικά εργαλεία. Αντί να απαγορεύουμε ριζικά τις απορρίψεις, θα έλεγα να τις μειώσουμε σταδιακά και να επενδύουμε περισσότερο στην επιλεκτικότητα, στην επιλεκτική αλλίευση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να σταματήσει την χρηματοδότηση της διάλυσης ε, των σκαφών. Έτσι όμως, ε, ίσως παραμείνουν σε ε, χρήση κάποια πεπαλαιωμένα σκάφη. Θα πρέπει να διατηρηθεί η ενίσχυση στη διάλυση σε συγκεκριμένε περιπτώσει, ώστε να μπορεί ένα ιδιοκτήτη παλιού σκάφου να επενδύσει σε ένα νέο σκάφο που θα τηρεί του περιβαλλοντικού κανόνε και του κανόνε ασφάλεια. Ε, Επίση, ε, θα μπορεί να επενδύσει σε ένα πιο ε, οικονομικό από, ενέργειας, από άποψη ενέργεια σκάφος πιο αποτελεσματικό, χωρίς να αυξάνει όμως την πλονάζουσα ε, χωρίς να αυξάνει την ελευτική του προσπάθεια. Επίσης, ε, λυπούμε που το ΕΤΘΑ δεν προβλέπει καμία ε, στήριξη των επαγγελματιών που υποχρεούνται να σταματήσουν προσωρινά τις δραστηριότητες τους για περίπτωση βιολογικής ανάπαυλας, σημαντικού ατυχήματος ή δυσμενών καιρικών συνθηκών. Εγώ προτιμώ στη, να στηρίξουμε τους επαγγελματίες ε, σε περίπτωση προσωρινής, προσωρινής παύσης των δραστηριοτήτων τους. Ό,τι αφορά την, ε, τη σταδιακή αύξηση των τιμών καυσίμων και ε, τη σημαντική επίπτωση στην αλία. Είμαι υπέρ προσωρινού μηχανισμού ε, της συγκυριακής ανόδου της τιμής του πετρελαίου προκειμένου να προφυλαχθούν οι, οι από απότομη ανόδου της τιμής του πετρελαίου σε ό,τι αφορά τι επενδύσει στα λιμάνια. Το άρθρο 41 αφορά επενδύσει στα ελληνικά λιμάνια πρωτίστω με σκοπό να υπάρξει διαχείριση των ανεπιθύμητων αλλιευμάτων. Δεν, άλλα, δεν προβλέπονται άλλα είδη επενδύσεων που είναι απαραίτητα για ανταγωνιστικά λιμάνια και τι ηχθιόσκαλες. Επιθυμώ διεύρυνση του πεδίου εφαρμογή του άρθρου 41, ώστε να μπορέσουν να υπάρξουν επενδύσει στο σύνολο των υποδομών των υφισταμένων λιμανιών. Το άρθρο 70 πλαισιώνει τη στήριξη τη αποθεματοποίηση. Προβλέπει ότι αυτή η στήριξη πρέπει να είναι ευθύνουσα έω την τελική της κατάργηση Το άρθρο 70 πλαισιώνει τη στήριξη της αποθεματοποίησης. Προβλέπει ότι αυτή η στήριξη πρέπει να είναι ευθύνουσα έως την κατάργησή της ε, το 2018. 19, συγγνώμη. Είμαι αντίθετο σε αυτή την προγραμματισμένη κατάργηση τη ενίσχυση τη αποθεματοποίηση και επιθυμώ να διατηρηθεί αυτό το σημαντικό εργαλείο για τη ρύθμιση τη αγορά προϊόντων αλληλεία. Αυτό το σύστημα επιτρέπει κατά κύριο λόγο να διασφαλίσετε η πώληση των προϊόντων σε συμφέρουσα για τους παραγωγούς τιμή. Σε ό,τι αφορά την υδατοκαλλιέργεια, χαίρομαι για τις φιλόδοξες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ό,τι αφορά την ε, βιώσιμη ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργεια, παρόλο που, όπως είπε ο κύριος Ρωμέβα το πρωί, θα πρέπει να μας γίνει και έμονη ιδέα. Είναι σημαντική η υδατοκαλλιέργεια, αλλά δεν θα πρέπει να μας γίνει και η ιδεολειψία. Το ΕΤΘΑ θα παρεμβαίνει για την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα, το ανθρώπινο κεφάλαιο, την περιβαλλοντική προστασία, τη δημόσια υγεία και την ασφάλιση των αποθεμάτων υδατοκαλλιέργεια. Σα υπενθυμίζω ότι η υδατοκαλλιέργεια θα, δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως αντίπαλο, αλλά ως συμπλήρωμα των αλληλευτικών δραστηριοτήτων επικροτώ τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, για την βιώσιμη και αλληλέγγυα περιφερειακή ανάπτυξη των αλληλευτικών περιοχών. Και μάλιστα, οι στρατηγικέ ολοκληρωμένη τοπική ανάπτυξη θα εφαρμοστούν από τοπικέ ομάδε δράση αλληλεία που εκπροσωπούν του διάφορου εμπλεκόμενου τομεί. Τα μέτρα, ολοκληρωμένα μέτρα ε, ε, τέτοια ανάπτυξη θα εφαρμοστούν από τοπικέ ομάδε με εμπλεκόμενου φορεί και θα ήθελα οι τομεί αλληλεία και τη να χαίρουν πλειοψηφική εκπροσώπηση σε αυτέ τι τοπικέ ομάδε δράσης αλληλείας. Ό,τι αφορά την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική. Η Επιτροπή προτείνει η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική να αποτελεί ένα απόσπαστο μέρο του ΕΤΘΑ, λαμβάνοντα τη μορφή τη άμεση διαχείριση. Για το σκοπό αυτό το ΕΤΘΑ θα χρηματοδοτήσει τη δικτύωση, το συντονισμό και τη συνεργασία, τι ανταλλαγέ καλών πρακτικών και τη βελτίωση των γνώσεων στον τομέα τη θάλασσα. Η Επιτροπή προτείνει τη χρηματοδότηση με 432 εκατομμύρια ευρώ για το χρονικό διάστημα 2014-2020 για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική. Κατά μέσο όρο ετησίω αντιστοιχεί το ποσό αυτό σε τετραπλάσιο περίπου το σημερινό προπολογισμό αυτή τη πολιτική η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική θα πρέπει να χαίρει επαρκού προπολογισμού, αλλά να μην γίνεται αυτό ει βάρος τη αλληλεία και τη υδατοκαλλιέργεια. Ενδείκνεται να αναλυθούν σε βάθο οι δημοσιονομικέ προτάσει τη Επιτροπής και ενδεχομένω να, θεσπιστεί ο καθορισμός ανώτατου ποσοστού του ΕΤΘΑ για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική. Αγαπητοί συνάδελφοι, λυπάμαι που μίλησα λίγο γρήγορα στην αρχή, αλλά όπως καταλάβατε θέλω τα ταμείο φιλόδοξο για να επενδύσει στο μέλλον της ε, Ευρωπαϊκής Αλίας. Δεν θα πρέπει να γίνει ένα μέσο επαναπροσανατολισμού επαγγελματικού των αλλιέων. πρέπει να είναι ένα μηχανισμός, ένα ταμείο που θα στηρίζει την αλία και τους αλλείς Περιμένω λοιπόν τις προτάσεις για τον κανονισμό αυτό και φυσικά είμαι στη διάθεσή σας και στη διάθεση των σχεδόν εισηγητών. Εννοείται για τα σχόλια και τις συζητήσεις και περιμένω με μεγάλο ενδιαφέρον τις τροπολογίες. Το χρονοδιάγραμμα το γνωρίζετε. 24 Σεπτεμβρίου, λίγη προθεσμία για την κατάθεση των, των τροπολογιών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κύριε Καντέκ. Θα δώσω το λόγο σε 7 ομιλητές που το ζήτησαν, 2-3 λεπτά το πολύ, ε, ξεκινώντας από τον κύριο Χάλαν. Ευχαριστούμε πολύ και ευχαριστούμε και για το έγγραφο εργασία. Είναι καλή αφετηρία για τι συζητήσει μα. Στο έγγραφο αυτό υπάρχουν πολλά πράγματα με τα οποία συμφωνώ. Υπάρχουν ορισμένα ζητήματα που χρήζουν ακόμα συζητήσεων και θα προσπαθήσω να τα αναφέρω. Θα ήθελα επίση να αναφερθώ σύντομα σε αυτά που είπε η Αμερικανίδα καλεσμένη μα, μας, ότι οι Αμερικανοί βρίσκονταν στην ίδια θέση που είμαστε και εμεί τώρα, ορισμένα χρόνια πριν, όταν είχαν υπεραλλιεύσει τα ήχθη θέματά του και έκαναν ένα φιλόδοξο σχέδιο, έθεσαν φιλόδοξου στόχου, έκαναν πολύ καλή δουλειά, άλλαξαν τα πράγματα και τώρα δεν έχουν τις ίδιες ε, προκλήσεις που έχουμε εμείς να αντιμετωπίσουμε με την υπεραλίευση έχουν ληφθεί μέτρα και βλέπουμε ε, με το παράδειγμα των Αμερικανών ότι τα μέτρα έπιασαν. Η έκθεση από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία των ΗΠΑ έδειξε ότι κατάφεραν να δημιουργήσουν μισό εκατομμύριο νέες θέσεις εργασίας με την λήψη των κατάλληλων μέτρων για την βιώσιμη ε, αλία και για την επιστροφή των ηχθιαποθεμάτων σε βιώσιμα ε, επίπεδα και κατάφεραν να κερδίσουν ένα δισεκατομμύριο με αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντική λοιπόν αυτή η έκθεση. Όσον αφορά τώρα αυτή την έκθεση, χαίρομαι πάρα πολύ που ο εισηγητής ε, καλεί για έναν ξαφή της ε, αλληλευτική ικανότητα και πιστεύω πως όλοι συμφωνούμε ότι χρειάζεται αυτός ο σαφή ορισμό Να τονίσω ότι οι Μαρικανοί ε, ορίζουν την ε, πλεονάζουσα αλληλευτική ικανότητα σε άμεση συνάρτηση με την υπεραλίευση. Όπου υπάρχει υπεραλίευση υπάρχει και πλεονάζουσα ικανότητα και ίσως αυτό απλοποιεί τα πράγματα, όμω υπονοεί ότι ίσω και εμεί να έχουμε πρόβλημα πλεονάζουσα αλληλευτική ικανότητα. Ε, εφόσον όλα μας τα ψάρια υπεραλλιεύονται και χρειάζεται να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα. Γι' αυτό λοιπόν προσωπικά τονίζω ότι δεν νομίζω ότι το ισχύον σύστημα είναι αρκετό για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα. Θέλουμε μια πιο μακροπρόθεσμη προσέγγιση και αυτό μου λείπει από αυτή την έκθεση. Τώρα όσον αφορά τις EFCs, πιστεύω πως συμφωνούμε ότι δεν μπορούμε να το θεωρούμε μόνη λύση υποχρεωτικό είναι όμως ένα μέτρο, είναι μία από τις επιλογές μας. Επίσης, χαίρομαι πολύ που ο κύριος Καντέκ τόνισε όσον αφορά την διαχείριση στόλου και ηχθιαποθεμάτων ότι χρειάζεται βελτίωση, χρειαζόμαστε βελτίωση στον τεχνικό εξοπλισμό και επίσης άλλο ένα θετικό είναι το ότι μπορεί να συζητηθεί το ζήτημα της σχετικής σταθερότητας και να ενθαρρυνθούν τα κράτη-μέλη να αναλάβουν το δικό τους μερίδιο της ευθύνης. Υπάρχουν λοιπόν αρκετά πράγματα με τα οποία συμφωνώ, είναι και εύκολο άλλωστε. Όσον αφορά επίση την έκθεση θα ήθελα να τονίσω ότι καλώς αναφέρατε την αρχή της ε, μέγιστη βιώσιμης απόδοσης με θετικό τρόπο. Επίσης, στην παράγραφο 3.1 τονίσατε το γεγονός ότι χρειαζόμαστε μια νέα γενιά αλλιέων. Και αυτό είναι καλό. Μετά στην παράγραφο 3.2 για τον εξυγχρονισμό και την ανανέωση του στόλου. Φυσικά βλέπω την ανάγκη ότι ε, πρέπει να συζητήσουμε περισσότερο για την ανανέωση του στόλου και αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει πόλο νέων επενδύσεων. Αλλά πρέπει να προσέξουμε τι θα γίνει με την χωρητικότητα, διότι έχουμε πολλέ περιπτώσει ανανέωση του στόλου με, ε, όπου διαπιστώθηκε πλεονάζουσα αλληλευτική ικανότητα. Θέλουμε λοιπόν λίγη προσοχή στι επενδύσει. Δεν ξέρω αν αυτέ οι, προ... οι επενδύσει θα επιφέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Σχετικά με την διάλυση των σκαφών. Νομίζω το ελεκτικό συνέδριο υπέβαλε μια έκθεση η οποία, σύμφωνα με την οποία το σχέδιο αυτό διάλυση δεν λειτουργεί έτσι όπως θα έπρεπε σε, όλα, σε όλους τους τομείς. Και σύντομα, Πρόεδρε, τελειώνω. Μάλλον, ας, θα τελειώσω εδώ, αφόσον θεωρείτε πως δεν έχουμε χρόνο. Νομίζω πως ανέφερα τα πιο σημαντικά. Ευχαριστώ. Ε, ε, ξεκινάμε λίγο καθυστερημένα επειδή δεν φτάνουν εγκαίρως οι ευρωβουλευτέ. Λοιπόν, ή προτείνω να ξεκινάμε λίγο αργότερα και μετά να βιαζόμαστε ή να τελειώνουμε λίγο αργότερα ή να ξεκινάμε εγκαίρως ακόμη και όταν έχουμε ένα βουλευτή στην αίθουσα. Αλλά δεν μπορούμε και να φτάνουμε καθυστερημένα και να μιλάμε όσο θέλει ο καθένας. Ο κύριος Ρωμέβα. Με συγχωρείτε αν άργησα κάπως. Όμως ε, έχασα απλώς το πρώτο μέρος της παρέμβασής σου. Να σε ευχαριστήσω λοιπόν. Γιατί πραγματικά πρέπει να εργαστούμε επί του κειμένου που μας έχει υποβάλει. Είναι ιδέες που ακολουθούν την κατεύθυνση που ήδη έχουμε συζητήσει. Με μερικά συμφωνούμε όπως την εξάλληψη του κεφαλαίου για τις μεταβιβάσιμες άδειες. Αυτό όντως πρέπει να το επιδιώξουμε. Και κάτι ακόμη πρέπει να επεξεργαστούμε, τον ορισμό της ικανότητας. Συμφωνούμε, πρέπει να το δούμε αυτό. Ο κύριος Χάγκλαντ μας έκανε μια πρόταση και εμείς θα κάνουμε κάτι ανάλογο. Αλλά δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να λέμε ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί πλέον ικανότητα χωρίς να ξέρουμε τι εννοούμε. Πρέπει να βρούμε έναν ορισμό που να είναι συνεκτικός και εφαρμόσιμος. Τώρα, να κάνω και εγώ κάποιες παρατηρήσεις για τις ποσότητες. Οι ποσότητες ορίζουν και τις προτεραιότητες. Το είπα και το πρωί. Θα θέλαμε εδώ να δείξουμε ότι ανησυχούμε για το γεγονός ότι γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια για έναν τομέα αυτών της υδατοκαλλιέργειας που δεν μπορεί να είναι λύση για τη σημερινή κατάσταση, ενώ από την άλλη λείπει. Η έμφαση που θα πρέπει να δίνεται σε άλλους τομείς. Και έπειτα υπάρχει το θέμα του ελέγχου. Αυτά είναι μεγάλα κεφάλαια στα οποία πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή. Στο ίδιο επίπεδο θα θέλαμε να αποφύγουμε. Να υπάρξει κακή χρήση των πόρων λόγω αύξησης των ικανοτήτων, ακόμη και αν το ονομάσουμε τελικά διαφορετικά. Ίσως το πρόβλημα να μην είναι η ίδια η ικανότητα, αλλά η βελτίωση. aussi la possibilité de pêcher euh, plus mieux. Εδώ λοιπόν υπάρχουν κάποιες πτυχές ότι, όπου θα πρέπει να, βελτιωθεί κάπως η διατύπωση και θα κάνουμε σχετικά κάποιες τροπολογίες, θα υποβάλουμε κάποιες τροπολογίες. Μια συγκεκριμένη πτυχή. Για την ε, αρχή της πρόληψης. Βάσει επιστημονικών γνώσεων θα πρέπει να υπάρξει εδώ η σωστή κατανομή. Και με την άδεια του Προέδρου εδώ να πω ότι υπάρχουν κάποια σημεία που λένε ότι μπορεί να χρηματοδοτούνται ενέργειες χωρίς εμπορικό όφελος. Εδώ υπάρχουν σίγουρα κάποιε πτυχέ που θα πρέπει να επεξεργαστούμε περαιτέρω και βάσει των τροπολογιών μα θα το επιδιώξουμε. Ευχαριστούμε κύριε Ρωμέβα. Κύριε Γκάλαχερ. Δύο παρατηρήσεις πρόεδρε. Το είπα προηγουμένω, αλλά δεν ήταν εδώ ο κύριο Κάντεκ. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται σε παραλληλισμό στην κοινή αλληλευτική πολιτική και την κοινή διακρατική πολιτική υπάρχει ένα συγκεκριμένο ποσοστό και ποσό το οποίο έχει απομονωθεί, θα αποδοθεί σε συγκεκριμένα ηγετικά προγράμματα. Εδώ θα πρέπει κύριε Καντέκ να δώσουμε έμφαση στην ε, ανανέωση μικρών λιμένων. Κάποιες φορές τα μεγαλύτερα σκάφη που αλλιεύουν τις ποσοστώσεις δεν μπορούν καθόλου να εκφορτώσουν εκεί. Θα πρέπει λοιπόν αυτές τις ε, τις εγκαταστάσεις που έχουν σχέση με τη θάλασσα να τις ενισχύσουμε. Το 94-95 η κυρία Φράγκα ήταν ήδη εδώ. Είχαμε ένα πρόγραμμα προώρησης ταξιδότησης για τους αλληλείς. Τώρα μιλάμε για μια νέα γενιά, ψαράδων. Δεν είναι τόσο χειρανακτική η εργασία τους βέβαια πλέον, αλλά να σκεφτούμε και αυτούς που εργάζονται σε δυσχερείς συνθήκες. Είναι χειρόνακτες. Και να σκεφτούμε εάν μπορεί να προβλεφθούν κονδύλια και για αυτούς τους ανθρώπους. Στα 55 οι περισσότεροι ε, αναγκάζονται να φύγουν από τη δουλειά. Εδώ όμως, αν θέλουμε να επιμεκίνουμε τον επαγγελματικό βίο, θα πρέπει να σκεφτούμε πώ θα του ενισχύσουμε και να δούμε ποια από τα μέτρα τη κοινή εργατική πολιτική μπορούμε να υλοποιήσουμε και στην ε, πολιτική αλία. κυρία Λόβεν. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ τον Αλέν Καντέκ για το έγγραφο εργασία. Ο συνάδελφο Ραούλ ε, ήδη ανέφερε τα σημεία με τα οποία συμφωνούμε. Εγώ θα μιλήσω περισσότερο για τα σημεία με τα οποία διαφωνούμε. Το είπα και το πρωί, κάποια στιγμή που χρειάστηκε και να φύγει, ότι βρισκόμαστε εν μέσω τη οικονομική κρίση. Και γίνονται έντονε συζητήσει στα κράτη-μέλη και στη δική μου πατρίδα ότι τα περισσότερα κονδύλια της Ένωσης θα πρέπει να πάνε σε καινοτομία και έρευνα και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Δεν υπάρχει ανοχή για τη χρησιμοποίηση κονδυλίων για παλαιομοδίτικο τρόπο χορηγήσεις, επιδοτήσεων σε γεωργούς, σε ψαράδες και ούτω καθεξής. Οπότε το γενικό μου σχόλιο είναι το εξής. Ακούσαμε και τα σχόλια της κυρίας Λουψέγκο από τις ΗΠΑ. Θα πρέπει να έχουμε τα μάτια μας καρφωμένα στο μέλλον και στο μέλλον θα πρέπει να ανακτήσουμε τα ελευτικά αποθέματα για να φτάσουμε σε επίπεδα μέγιστης βιώσιμης απόδοσης. Οι επιστημονικές μελέτες δείχνουν ότι αν έχουμε αποθέματα άνω της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης θα αυξηθούν και οι θέσεις εργασίας, θα αυξηθεί η αλίευση και θα αυξηθεί και το κέρδος και για τον αλλιευτικό κλάδο. Φοβάμαι ότι το εγγράφο εργασία σας παρά είναι προσανατολισμένη στην παρούσα κατάσταση Εκεί χρειαζόμαστε οικονομική στήριξη για τον εξυγχρονισμό του στόλου, για την κατασκευή νέων σκαφών. Και η πρότασή σας για χορήγηση από επιδοτήσεων διάλυσης και τη χρησιμοποίηση των κονδυλίων ε, για να κατασκευαστεί νέο πλοίο, το κονδυλίο διάλυσης και την κατασκευή νέων πλοίων, είναι κάπως επιχειωμένες αυτές οι προτάσεις όπως ε, καταλαβαίνουν οι μικροί επιχειρηματίες, για να μπορέσουν να επενδύσουν στο μέλλον θα πρέπει πρώτα να κερδίζουν, να βγάζουν τα ζήν, μόνοι τους, να μην εξαρτώνται από κανέναν. Και αν θέλουμε να ε, αποκαταστήσουμε τα ηχθή αποθέματα, θα πρέπει αυτό να το έχουμε υπόψη. Δεν συμφωνώ με την επαναφορά των επιδοτήσεων διάλυσης, επιδοτήσεων αποθεματοποίησης, εξυγχρονισμού, επιχορηγήσεων για τα καύσιμα εγώ είμαι αισιόδοξη και πιστεύω ότι ο κλάδος κλάδο οι ψαράδε θα καταφέρουν να βγάζουν από μόνοι του τα προ το ζήν, χωρί να χρειάζονται τι δικέ μα επιδοτήσει. Ελπίζω να συνεχίσουμε τις συζητήσει στην Επιτροπή μας και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να δούμε αν μπορούμε κάπως να συνεννοηθούμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Λόβεν, κυρία Ντότζ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομα σχόλια για το σημείο αυτό. Ευχαριστώ τον Αλάν Καντέκ για την έκθεσή του. Είμαι στην ευχάριστη θέση να συμφωνώ με ένα μεγάλο τμήμα του γράφου εργασία και των όσων μα είπε. Έχω κάποιε ανησυχίε για το θέμα τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση και τη δυνατότητα να επιτύχουμε τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση σε όλα τα διεχθεία αποθέματα ταυτόχρονα στην κοινή πολιτική. Νομίζω ότι αυτό το σημείο θα πρέπει περαιτέρω να το δουλέψουμε. Ένα από τα σημεία που με ικανοποιούν είναι ο τόνος, το ύφος ε, της έκθεσης αυτής του εγγράφου εργασίας. Μερικές φορές η Αλληλευτική Επιτροπή μιλά με καταθλιπτικό τρόπο για τον απειρχιωμένο στόλο, για τη σπάνη των αλληλευτικών αποθεμάτων. Όλα αυτά είναι κάπως ζωφερά και αποκαρδιωτικά. Όπως είπε και η Ζαμπέλ, στο μέλλον θέλουμε μια αλία που θα είναι και βιώσιμη και ανταγωνιστική και το ύφο όλων αυτών που λέμε, το, ο τόνος όλων αυτών που κάνουμε, είναι σημαντικό. Θα πρέπει να φαίνεται από τον τόνο της, ε, των προτάσεών μα και από το ύφο μια αισιοδοξία για να περάσει αυτό το μήνυμα και στους ψαράδε και στι αλληλευτικέ κοινότητε γενικώ. Τώρα το θέμα της πλεονάζουσας αλληλευτική ικανότητας και το θέμα του ορισμού τη. Θα το εξετάσουμε και επ' ευκαιρία της έκθεσης Ροντάστ θα πρέπει πρώτα να συμφωνήσουμε τι εννοούμε με την ε, πλεονάζουσα αλληλευτική ικανότητα. Τον αριθμό των αλληλευτικών σκαφών ε, εννοούμε. Εννοούμε στη, το συγκεκριμένο αριθμό σκαφών, αλλά την δυνατότητα αλλήλευσης συγκεκριμένου αριθμού ψαριών. Θα πρέπει να ορίσουμε με σαφήνεια την, την αλλιευτική ικανότητα και επίση να λάβουμε υπόψη και την αλληλεία μικρή κλίμακος και τι παράκτιε κοινότητε που έχουν περιορισμένες εμβέλειες αλλιεία. Εκεί η ικανότητα μειώθηκε σταδιακά, όπω στη Βόρεια Ιρλανδία για παράδειγμα, από όπου κατάγομαι. Εκεί είχαμε αισθητή μείωση τη αλλιευτική ικανότητα. Και μπορεί να έχουμε ένα-δυο μεγάλα σκάφη, τα οποία ισοδυναμούν την ικανότητα 20 μικρότερων και παλαιότερων σκαφών. Δεν θέλουμε να εξαλείψουμε την παράκτη αλία ή τραλία μικρή κλίμακο. Προσοχή! Γι' αυτό και θα πρέπει να είμαστε πολύ σαφεί και συγκεκριμένοι στι προτάσει μα. Πολύ φοβάμαι θα δημιουργηθεί πρόβλημα από αυτό το σημείο. Ο κύριο Γκάλεχερ μίλησε για τα μικρά λιμάνια. Συμφωνώ, συμφωνώ. Είναι το θέμα ευαίσθητο και στη δική μου εκλογική περιφέρεια. Έχουμε πολύ μικρά λιμάνια που δεν μπορούν, δεν μπορούν να ελιμενιστούν σκάφη γιατί θα πρέπει να γίνουν κάποιες εργασίες λόγω της περιορισμένης ικανότητας. Ευχαριστούμε κυρία Τότση, κυρία Ρόντουστ. Και εγώ θα είμαι σύντομη. Καταρχάς, να ευχαριστήσω για την έκθεση. Κάποια πράγματα τα υποστηρίζω χωρίς δεύτερη σκέψη. Και τώρα θα επικεντρωθώ όμω σε αυτά με τα οποία διαφωνώ. Εάν θέλουμε να έχουμε ψάρια που θα μας δίνουν ένα καλό εισόδημα, πρέπει πραγματικά να δούμε εάν υπάρχουν αρκετά ψάρια στις θάλασσές μας, εάν μπορούμε να το διασφαλίσουμε. Και γεγονός είναι ότι πολλά από τα ψάρια έχουν υπεραλλιευθεί. Εάν θεωρήσουμε τον ψαρά ως επιχειρηματία, τότε για μένα αυτό σημαίνει ότι πρώτα πρέπει να πάει στην τράπεζα και να αποδείξει ότι η επιχείρησή του τρέχει τόσο καλά, ότι έχει τόσο τζίρο, τα τελευταία 10 χρόνια μπορεί, θα μπορέ, τα, επόμενα 10 χρόνια θα μπορέσει να τρέξει καλά την επιχείρησή του και μετά η τράπεζα να του δώσει το χρηματικό ποσό που χρειάζεται. Με την προϋπόθεση ότι θα μπορέσει φυσικά να πληρώσει και τις οφειλές του. Οι τράπεζες όμως αυτό δεν το κάνουν και δεν το κάνουν γιατί νομίζουν πως έχουμε αρκετά ψάρια δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια μας σε αυτό το πράγμα. Σε ορισμένους τομείς έχουμε πάρα πολλά πλοία και πολύ λίγα ψάρια. Και πώς θα αντιστρέψουμε την κατάσταση. Πρέπει να φροντίσουμε στους τομείς αυτούς να έχουμε λιγότερα πλοία. Γι' αυτό λοιπόν και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν κάνουμε ε, λόγο για ε, πλεονάζουσα λευτική ικανότητα. Ε, φυσικά και την έχουμε. Την έχουμε εκεί στις περιπτώσεις όπου οι άνθρωποι δεν τηρούν τις ποσοστώσεις. Και έχουμε τέτοιες περιοχές στην Ευρώπη, φυσικά και το ξέρουμε, όλοι το ξέρουμε. Εάν όλοι οι ψαράδες τηρούσαν τις ποσοστώσεις, δεν είχαμε καμία ανάγκη να βρισκόμαστε εδώ σήμερα. Ναι, οκ, και δεν χρειαζόμαστε λοιπόν και αυτές τις ε, διατάξεις. Ξανά θα το πω, θέλουμε δεδομένα. Χρειαζόμαστε επιστημονικά δεδομένα και, και χρειάζεται να δούμε πώς τα ψάρια θα έχουν ικανοποιητικούς αριθμούς, οι αλληλείς θα μπορέσουν να, να χρηματοδοτηθούν από τις τράπεζες κτλ. Τώρα, όσον αφορά τον στόλο, είμαι υπέρ της χρηματοδότησης του στόλου, εάν όμως μπορέσουν να αποδείξουν ότι δεν έχουν πλέον πλεονάζουσα αλληλευτική ικανότητα, εάν ε, καταφέρουν να αποδείξουν ότι όλα είναι σύμφωνα με, τα προβλεπόμενα και εάν μπορέσουμε να, να διασφαλίσουμε ότι η, μικρή, η αλληλεία μικρής κλίμακας και η παράκτια αλληλεία τα επόμενα χρόνια θα μπορέσει να επιβιώσει σε και να διατηρηθεί σε βιώσιμα επίπεδα. Για όσο δεν μπορούμε να το διασφαλίσουμε αυτό, θα συνεχίσουμε να έχουμε να υπάρχουν ανησυχίες, θα συνεχίσουμε να έχουμε προβλήματα. Θα συνεχίσουν τα σύγχρονα αλλιευτικά σκάφη να υπεραλλιεύουν τα αποθέματα και αυτά τα αποθέματα θα συνεχίσουν να μειώνονται ακόμα περισσότερο από ότι τώρα. Για την ανανέωση του στόλου. Ναι, να το κάνουμε. Να το κάνουμε όμω εκεί που δεν υπάρχει πλεονάσια ελευτική δυνατότητα. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστούμε ο κύριος Ντέιβις. Μάλιστα. Νομίζω ότι ο κύριος Καντέτ ανήκει σε λάθος κοινοβουλευτική ομάδα. Θα έπρεπε να είναι στην ΚΟΕ. Όχι μόνο θέλει να καταργήσει τις ε, επιδοτήσεις, αλλά έχει και τα βλέπει όλα τόσο μαύρα. Είδατε πόσο θετική ήταν η κυρία Λουτσέγκο. Σωστα... Ε, μίλησε για σωστά μέτρα, για δύσκολου στόχου, να, να δούμε τη μέγιστη βιώσιμη απόδοξη, ε, απόδοση και μετά από όλα αυτά να ανακάμψουν οι πληθυσμοί των ψαριών και να δημιουργηθούν και νέες θέσει εργασίας. Έτσι, η θεώρηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας είναι μαύρη και άραχνη. Δύσκολα τα πράγματα στις αγορές, δύσκολα τα πράγματα με τα ηχθιαποθέματα. Δεν μπορούμε έτσι να δημιουργήσουμε μία κερδοφόρο αλληλευτική βιομηχανία, αν τα βλέπουμε όλα μαύρα. Δύο πράγματα θέλω να τονίσω. Καταρχάς, ο Κάρλ Χάγκλουν ότι δεν υπάρχει υπεραλίευση. Ή μάλλον ότι όπου υπάρχει υπεραλίευση υπάρχει και, μέγιστη και πλεονάζουσα δυνατότητα. Εγώ λέω, και επίσης μα είπε μάλλον ότι δεν έχει αποδειχθεί αυτό. Ε, ωραία, άμα δεν έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει πλεονάζουσα ικανότητα, τότε α καταργήσουμε τις ε, για τη διάλυση των σκαφών. Αυτό που λείπει από το έγγραφο αυτό, εφόσον δεν υπάρχει κάποια αναφορά στα, στα κεφάλαια που θα υπάρχουν στο Ταμείο, είναι Έχουμε επιδοτήσεις για την διάλυση, επιδοτήσεις για τα καύσιμα, επιδοτήσεις για όλες τις ε, υπάρχουσες υποδομές των λιμένων. Τι θα περικοπεί όμω για να πάνε τα χρήματα εκεί. Η Κομισιόν μας ε, παρουσίασε ορισμένε ιδέες με τις οποίες θα μπορέσουμε να υποστηρίξουμε τους ψαράδες, τις παράκτιες κοινωνίες, να βάλουμε τα χρήματα λοιπόν εκεί και πολλά από αυτά που εσείς υποστηρίζετε ε, δεν μας λένε από πού θα περικοπούν τα κεφάλαια για να πάνε εκεί. Ε, κυρία Μιράντα, ευχαριστώ. Θα είμαι αρκετά συνοπτική. Μπορούμε να μιλάμε ώρες ολόκληρες για, να, για το αν θα θέλουμε μέγιστη βιώσιμη απόδοση, αν θέλουμε λιγότερη περισσότερη οικολογική πολιτική, αλλά σε τελική ανάλυση, χωρίς ε, δείκτες, χωρίς στατιστικά στοιχεία, χωρίς δεδομένα είτε κοινωνικο-οικονομικά είτε περιβαλλοντικά, χωρίς μελέτες δεν θα έχουμε απαραίτητα στοιχεία για να καθορίσουμε τι είδου βιώσιμη αλία θέλουμε, αν θα είναι παράκτια ή ανοιχτή θάλασσα, ή βυθοπέλαγη και ούτω καθεξής. Εμείς θα καταθέσουμε τροπολογίες για τον επιστημονικό κλάδο και τις συνεργασίες επιστημονικών και λευτικών κλάδων. Νομίζω ότι χωρίς στοιχεία και χωρίς στατιστικές δεν έχουμε που να στηριχθούμε. Μπορούμε να μιλούμε γενικά και όριστα. Στο Βίγκο έχουμε την, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ελέγχου της Θάλασσας. Εκεί είναι σαφής η πρωτοβουλία για την θάλασσα με συνεργασία των επιστημόνων, των επιχειρηματιών, των αλλιέων και με συνεργασία με πανεπιστήμια της Βόρειας Πορτογαλίας και επιχειρηματίες της Βόρειας Πορτογαλίας. Πρόκειται για ένα πιλωτικό πρόγραμμα που μπορεί να έχει επιρροή και στην ολοκληρωμένη πολιτική θάλασσας, αλλά να συνδυαστεί και με τα καινοτόμα προγράμματα της στρατηγικής του 2020. Θα μπορούσε το οργανισμός του Βίγο να γίνει ένα είδος εργαστηρίου για αναλύσεις και μελέτες της, ε, θαλάσσιας, της ολοκληρωμένης θαλάσσης πολιτικής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μάλλον και εγώ λάθος θα κάνω, γιατί νόμιζα ότι στο Κοινοβούλιο εξετάζουμε ιδέες και προτάσεις μέσα σε ένα ε, ιδεολογικό πλαίσιο αναφοράς. Και δεν θα α, ε, αντικατοπτρίζουμε εδώ τις κομματικές ιδεολογίες κατά ανάγκη. Ευχαριστώ τον εισηγητή για τις θέσεις του και θα ήθελα να υποβάλω κάποιες παρατηρήσεις, να κάνω κάποιες συστάσεις και προτάσεις, πείτε τις όπως θέλετε. Γνωρίζουμε ότι το Ταμείο που έχει συγκεκριμένο προπολογισμό, θα αφιερώσει 1 δισεκατομμύριο 47 εκατομμύρια για την άμεση διαχείριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για ποιο λόγο όμω αυτή η άμεση διαχείριση. Και χάρη διαφάνεια θέλουμε να ξέρουμε πού θα αφιερωθούν αυτά τα κονδύλια, τι θα χρηματοδοτήσουν. Παρακαλώ να περιληφθεί αυτό στην έκθεση. Επίση, το ταμείο αυτό, το ΕΤΘΑ, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να συμβάλλει ε, στο στην προσαρμογή του κάθε λευτικού στόλου, εθνικού και τοπικού, στις οικονομικές συνθήκες, στις κοινωνικές, περιβαλλοντικές, αλλά και πολιτιστικές συνθήκες. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ε, είσοδο των νέων αλλιέων στον κλάδο, πολύ σημαντικό αυτό το θέμα, θα ήθελα να περιληφθούν κάποιες οικονομικές ενισχύσεις που θα περιλαμβάνουν και την οικονομική και εργασιακή αναγνώριση, αλλά και μισθολογική ε, αναγνώριση, καθώς και την προστασία των γυναικών που απασχολούνται στον κλάδο και που συμβάλλουν στην ανάπτυξη ε, της αλίας, της υδατοκαλλιέργειας και της οικονομίας γενικώ. Θα σας πρότεινα επίσης, σε ό,τι αφορά τις θεομηνίες ή φυσικές καταστροφές ή τον περιορισμό της βιομάζας, που μπορεί να οδηγήσει σε ακινητοποίηση, να δημιουργηθεί ένα ταμείο κρίσης, ε, αντιμετώπισης ε, κατεπηγόντων περιστατικών. Επίσης, ό,τι αφορά τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, ε, φαίνεται ότι οι Κανάρι νήσοι έχουν εξαφανιστεί από τη φετινή πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εγώ θα ήθελα να ξαναπεριληφθούν και να, περιληφθεί επίσης, να περιληφθούν επίσης και οι Βαλεαρίδες νήσοι, γιατί είναι αρχιπέλαγος. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις επιδοτήσεις για την προσαρμογή του ελευτικού στόλου και τις επιδοτήσεις για τη διάλυση των σκαφών, συμφωνώ ότι είναι ε, αμφισβητήσιμο το θέμα χωρίς να έχουμε επιστημονικά πορίσματα την ε, αλληλευτική ικανότητα. Οπότε θα πρέπει να διατηρήσουμε τις επιδοτήσεις διάλυσης και να ελέγξουμε ότι όντως χρησιμοποιούνται αυτές οι επιδοτήσεις για διάλυση και όχι για αύξηση της αλληλευτικής ικανότητας. Επίσης συμφωνώ με τον εξυγχρονισμό του στόχου γιατί έτσι θα εξασφαλίσουμε ε, υγιεινή, ε, περιβαλλοντική προστασία, περιορισμό διοξιδίου του άνθρακα, ενεργειακή ε, εξοικονόμηση, προστασία και ασφάλεια των αλλιέων και να προβλέψουμε μια ουσιαστική μεταρρυθμίση της αλληλευτικής πολιτικής με ελάχιστο προπολογισμό. Και τέλος, γιατί αμφισβητείτε τόσο το γεγονός ότι υπάρχουν επιδοτήσεις ή ενισχύσεις για τον αναπροσανατολισμό και ανασυγκρότηση ενός στρατηγικού κλάδου που ούτως ή άλλως ε, αποτελεί τμήμα όχι μόνο της οικονομίας αλλά και της διατροφής μας και δεν ε, αμφισβητούμε τις επιδοτήσεις στα αυτοκίνητα ή στα καύσιμα ή στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Γιατί ο καθένας... Ε, ε, προτάσει την ε, ιδεολογία του, αλλά τελικά θέλει να ε, συγκεντρώνει τις επιδοτήσεις στους κλάδους που ανθούν στη δική του πατρίδα. Στην Ισπανία τις μεταφιέσεις τις κάνουμε κυρίως στην εποχή του καρναβαλιού. Ο κύριος Μιλάνα. Πολύ σύντομα, και δεν έχουμε χρόνο. Α, με αφήνεις. Εντάξει, ευχαριστώ. Νομίζω ότι είχαμε μια ακρόαση το πρωί πολύ ενδιαφέρουσα. Ζητήσαμε απλούστευση, απλότητα και σαφήνεια. Η προσπάθεια λοιπόν που να κάνουμε είναι κατά κύριο λόγο στην κατεύθυνση της απλούστευσης και πρέπει να διευκρινίσουμε και εδώ και στην έκθεση για το βασικό κανονισμό τι είναι οι ικανότητε, τι είναι η μικρή κλίμακα αλίας και τι είναι ο ελευθερικός τουρισμός. Αυτά απαιτούν συγκεκριμένους, σαφείς, ορισμούς συνενετικού για το μέλλον. Διότι δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε αν δεν τα θέσουμε αυτά από την αρχή σωστά. Δεν θα πετύχουμε το στόχο μας. Συμφωνώ απολύτω με πράγματα που άκουσα από το πρωί για το ποσοστό συγχρηματοδότηση, για τη συλλογή δεδομένων, για την ε, στήριξη των δραστηριοτήτων ελέγχου. για την ε, βιολογική ή την, ε, την πάυση αναπεριοχή. Επίσης, για τους λιμένες θα πρέπει να υπάρχει χρηματοδότηση. Όμως, όταν η χρηματοδότηση έχει να κάνει με τη συντόμευση της απόστασης μεταξύ ψαρά και εμπορευμένου, δηλαδή εγκαταστάσεις που να προσφέρουν προστιθέμενη αξία στον τομέα της αλίας, αυτό να ενισχύεται. Όπως ε, για, την, ε, για τα κατεψυγμένα προϊόντα, την αποθήκευση. Όταν η παρέμβαση στο λιμάνι στηρίζει την αλληλευτική δραστηριότητα δηλαδή. Αυτό να χρηματοδοτείται. Όμως, σε σχέση με τον κύριο Ραού διαφέρει διαφέρει απόψη μου λίγο για την επατοκαλλιέργεια. Πρέπει να ξεφύγουμε από την ιδεολογική τοποθέτηση στο θέμα αυτό δεν επιλύει τα προβλήματα της αλίας ή το καλλιέργεια, αλλά των επιστημιστικών μας αναγκών. Αυτό είναι το ζητούμενο. Χρειαζόμαστε τρόφιμα και η παράνομη αλεία πολλές φορές σήμερα ακριβώς οφείλεται στις πολύ μεγάλες, στην πολύ μεγάλη ζήτηση που πιέζει στο χώρο αυτό. Στη Γεωργία τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Εγώ θέλω να υπάρχει βιολογική υδατοκαλλιέργεια που να σέβεται το περιβάλλον που να επιτρέπει την ανάλογη προστασία και τη συντήρηση. Όμως, γιατί συμβαίνει αυτό είναι άλλο θέμα. Είναι ένα φαινόμενο που υπάρχει και δεν μπορούμε να το αρνηθούμε. Η ζήτηση για τα ψάρια αυξάνεται παγκοσμίω. Εδώ λοιπόν υπάρχει σημαντική ζήτηση και πρέπει να δοθεί μια απάντηση. Εάν ακριβώς γιατί αυτή η ζήτηση είναι υπαρκτή, εάν με αυτήν απαντήσουμε σε πλεονάζουσα, με πλεονάζουσα ή παράνομη αλεία, τι σημαίνει αυτό. Όχι καν δεν θα επιλύσουμε, αλλά θα αφαιρέσουμε ένα μέρος των πόρων. Αυτό είναι το θέμα. Εγώ είμαι ανοιχτό στη συζήτηση αυτή. Δεν έχω προκαταλήψεις. Δεν είμαι υπέρ ούτε κατά. Και μια τελευταία παρατήρωση, Πρόεδρε, πολύ σύντομα. Για τι μεταβιβάσιμε άδειε, Αλία. Εδώ να πω ότι είμαι τελείω αντίθετο. αλλά όχι για τις ατομικές άδειες. Προσοχή. Πρέπει να κάνουμε μια διάκριση εδώ. Η κατεύθυνση του βασικού κανονισμού που θα πρέπει να συζητήσουμε και που τελικά δεν καταλήξαμε σε συμπέρασμα, τι μας λέει. Λέει όχι στη μεταβίβαση αδειών, αλλά ναι στις ε, ατομικές άδειες. Εάν αυτό είναι η κατάληξη, το Ταμείο δεν θα μπορεί να καλύψει αυτή την εξέλιξη. Ευχαριστούμε. Είχατε δίκιο, κύριε Καντέκ, δεν μπορούσατε να είστε σύντομο. Η κυρία Μπιλμπάου, θα προσπαθήσω να είμαι λακωνική σε ό,τι αφορά την έκθεση. Υπάρχει κάτι που λείπει από την έκθεση Καντέκ και είναι νευραλγικό θέμα. Φαίνεται ότι όλοι θέλουμε έναν προσωδοφόρο αλληλευτικό κλάδο. Οπότε από αυτό θα πρέπει να ξεκινήσουμε, από αυτή τη βάση, για να έχουμε μια προσοδοφόρα αλία. Τι θα πρέπει να κάνουμε στην Ευρώπη. Υπάρχει πλεονάζουσα ικανότητα. Ξέρουμε τον ορισμό, μικρές ποσοστώσεις, λίγο ψάρι. Αλλά το θέμα της πλεονάζουσας ικανότητας φαίνεται ότι διωγγώνεται. Υπάρχει μια υπερβολή. Οπότε, αν υπάρχει υπερβολή, θα πρέπει είτε να περιορίσουμε τον αριθμό των σκαφών, οι πρώτε επιτροπή είναι μεταβάσιμε σε ελληνικέ παραχωρήσει, ώστε με φυσικό τρόπο να συγκρατήσουμε τον κλάδο. Αν διαφωνούμε, θα πρέπει να έχουμε ένα σαφέ πρόγραμμα και να εφαρμόσουμε το πρόγραμμα τη διάλυση σκαφών. Δεν μπορούμε όμω να τα δεχόμαστε όλα. Το ενδιαφέρον στη συζήτηση και η προσπάθεια που θα πρέπει να κάνουμε είναι η εξή. Να δούμε τι έχουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν είναι δύσκολο να κάνουμε ένα απολογισμό. Βέβαια δεν έχουμε ούτε πολλά στοιχεία ούτε πολλές πληροφορίες. Την πρώτη μέρα που μας έκανε η κυρία Δαμανάκη η Επίτροπος την πρόταση, στην, ε, την πρόταση της στην Επιτροπή ελεία ήταν το μόνο πράγμα που τη ζήτησα. Πληροφορία, ενημέρωση για τον αριθμό των σκαφών. Πληροφορίες για την πιθανή ενδεχόμενη ε, πλεονάζουσα ικανότητα, για την πιθανή υπεραλίευση, ώστε τεκμηριωμένα να μπορούμε να κρίνουμε. Γιατί ο καθένα μπορεί να υποστηρίζει τη θέση του, αλλά ουσιαστικά μιλάμε χωρίς στοιχεία. Υπάρχουν χώρε και περιοχές που τα τελευταία 10-15 χρόνια εφάρμοσαν σημαντική ανασυγκρότηση του στόλου τους και μάλιστα ε, χειρίστηκαν και σωστά τα κονδύλια για τη διάλυση. Δεν φαίνεται όμως αυτό που θένα στην έκθεση. με την ανασυγκρότηση, παρά την ανασυγκρότηση που έκαναν θα πληρώνουν τα σπασμένα και των υπόλοιπων που δεν προέβησαν σε ανασυγκρότηση. Με όλη τη συζήτηση που κάνουμε και τις εύλογες θέσεις που έχουμε, λύση δεν βλέπω. Αν πούμε σε κάποιον, αυτή είναι η μεταρρύθμιση της κοινή ελευθερικής πολιτικής. Αυτό είναι το σχέδιο. Τόσα πλοία έχουμε, τόσα ελευθερική δυνατότητα, τέτοια ήχθη αποθέματα και αν κάνουμε τους λογαριασμούς θα δούμε ότι δεν βγαίνουν τα κουκιά. Δεν υπάρχουν αρκετά, αρκετά ψάρια για όλους. Θέλουμε όμως προσοδοφόρα αλεία. Αν θέλουμε προσοδοφόρα αλεία και υπάρχει ε, υπερβολική ε, ικανότητα και το γνωρίζει ο κλάδος, άρα κάτι θα πρέπει να γίνει. Ανασυγκρότηση με τον ένα ή τον άλλο τρόπο για τους νέους. Σιγά μην πάνε οι νέοι να ψαρέψουν αν δεν είναι κερδοφόρα επικερδής η αλεία. Θα πρέπει λοιπόν να εφαρμόσουμε τρόπους για να γίνει πιο επικερδής αυτή η αλληλευτική προσπάθεια, αυτή η αλληλευτική δυνατότητα. Μόνο έτσι θα καταφέρουμε να εφαρμόσουμε μια κοινή αλληλευτική πολιτική στην Ευρώπη. Αλλιώς, χωρίς στοιχεία, όσο και να συζητάμε και όσο, όσε θέσει και να έχουμε, τι μας αρέσει και τι δεν μας αρέσει, δεν υπάρχει υπόβαθρο και δεν υπάρχει σαφήνεια για το πως θα που οδεύομαι. Κύριε Καντέκ, παρακαλώ, συντομή, γιατί έχουμε και άλλο θέμα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κατά πρώτον, να ευχαριστήσω άπαντε. Για το πάθος και τον ενθουσιασμό <clears throat> με τα οποία τοποθετηθήκατε για το θέμα αυτό. Δείχνει ότι σας ενδιαφέρει ιδιαίτερο. Και μελετήσατε κιόλα την έκθεση. Δεν θα απαντήσω στον καθένα ξεχωριστά θα τα ξανασυζητήσουμε. Απλώς να σας πω ότι υπολογίζω σε εσά για τη συνεργασία σας, τις τροπολογίες σας, για να συζητήσουμε διμερώς με τους ΜΕΝ και του ΔΕ και να προχωρήσει το όλο θέμα μαζί με τον βασικό κανονισμό. Απλώς μια σύντομη παρατήρηση κατά ότι η πλειοψηφία από εσά θεωρεί ότι πρέπει επιτέλους να ορίσουμε την ικανότητα και την υπεραλίευση. Νομίζω η πλειοψηφία έτσι, όχι όλοι, να απαντήσω σε κάποιον από εσά, έναν και μόνο, που απευθύνθηκε σε μένα προσωπικά, τον κύριο Ντέβις δηλαδή. Ε, κύριε συνάδελφε, υπερβάλλετε λίγο, ως συνήθως. Το έχουμε συνηθίσει βέβαια, έτσι. Σας διαβεβαιώ λοιπόν. Εάν αυτό σας καθησυχάζει. Δεν είμαι εκλεγμένος της άκρας αριστεράς, είμαι από τη δεξιά παράταση και αναλαμβάνω την ευθύνη. Δεν είμαι ε, ακραίος φιλελεύθερος, αυτό είναι θέμα ζούγκλας, αλλά ως φιλελεύθερος πιστεύω στην ελευθερία. Ας είμαστε λοιπόν σαφείς. Δεν σημαίνει ότι επειδή κάνω τέτοιες προτάσεις είμαι ακροαριστερός και τα θέματα αυτά δεν έχουν καθόλου πολιτική διάσταση και κομματική, αλλά διαπαραταξιακή. Θα πρέπει λοιπόν να μην είμαστε εδώ δημαγωγοί στην προσέγγιση μας. Αυτό θα το κάνουν οι κομματικοί θύνοντες στα διάφορα κράτη-μέλη. Τώρα, για τις συγκεκριμένε προτάσεις που έχω αποβάλει, είναι προτάσεις... Γι' αυτό έτσι ονομάζονται, γι' αυτό και πρόκειται να τις συζητήσουμε και γι' αυτό μιλούμε για τη χρηματοδότηση προτινόμενων μέτρων. Πρέπει να τα συζητήσουμε. Βεβαίως, το, το ταμείο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Θάλασσα και την Αλία διαθέτει 6,5 δι. Δεν διαθέτει ούτε παραπάνω ούτε λιγότερα. Αυτά θα πρέπει να διαθέσουμε και αυτά θα πρέπει να αποφασίσουμε. Αυτά ήθελα να πω, Πρόεδρε. Νομίζω ότι έχουμε ευκαιρία να τα ξανασυζητήσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Καντάκη και περάμε στο τελευταίο σημείο τη ημερήσια διάταξη για σήμερα. Τι ε, κοινέ διατάξει για τα Ευρωπαϊκά Ταμεία και κατάργηση του κανονισμού 1083 του 2006. 20 λεπτά μα έχουν μείνει για την εξέταση και τη συζήτηση. Παρακαλώ, ποιοι θα λάβουν το λόγο στη συζήτηση για να υπολογίσω πόσο χρόνο δικαιούται ο καθένας. Το λόγο έχει ο κύριος Ζαν Πολ Μπεσέ για να μας παρουσιάσει το σχέδιο γνωμοδότησής του. Θα είμαι πολύ σύντομος, Πρόεδρε, διότι η όλη η συζήτηση, η, επί της συζήτηση, έχει ήδη γίνει με την αφορμή τη της του κυρίου Καντέκ για το Ταμείο της Θάλασσας και της Αλίας. Εδώ, όπως είχα πει και στην προηγούμενη συνεδρίασή μας, θέλω απλώς να τοποθετηθώ για το συνολικό κανονισμό, για όλα τα ταμεία και για τις γενικές αρχές που θα τα διέπουν. Εδώ θα πρέπει να οργανώσουμε την κατανομή όλων των ευρωπαϊκών κονδυλίων, εκ των οποίων μέρος αποτελεί η Αλία. Το ο γενικός αυτό κανονισμό, όπω είχα πει και την περασμένη φορά, είναι ένα εργαλείο που πιστεύουμε ότι έχει τοποθετηθεί σε ένα θετικό πλαίσιο, διότι επιτρέπει τη μεγαλύτερη συνεκτικότητα των πολιτών, υπάρχει διάθεση εναρμόνισης και μεγαλύτερη αιρεσιμότητα σε σχέση με τους στόχους των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδίω ό,τι αφορά την βιωσιμότητα των πόρων και το θέμα των κλιματολογικών συνθήκων. Εδώ επιτρέπεται για καλύτερη εδαφική προσέγγιση και ενίσχυση των ε, τοπικών ε, αρμοδιοτήτων. Κάτι που νομίζω ότι σε όλους μας είναι προσφυλές. Σε ό,τι αφορά τον ίδιο τον τομέα της αλίας, ο γενικός αυτός κανονισμός στις γενικές του αρχές δεν ε, παρουσιάζει διάθεση επαναχώρησης ή νέους φραγμούς όλες οι νέες αρχές και οι νέες ρυθμίσεις ευνοούν την θέσπιση μιας νέας αλληλεκτικής πολιτικής με ένα καινούργιο προσανατολισμό της βιώσιμότητας ε, των ε, πόρων και των θέσεων εργασίας. Εδώ θέλω να σταθώ σε τρία συγκεκριμένα σημεία. Το πρώτο, τροπολογία επαριθμών 1, ευρύτερη εφαρμογή της έννοιας της επικουρικότητας προκειμένου να ισχύει και για τους δικαιούχους μικρού όγκου που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλίας. Δεύτερη τροπολογία που εντοπίζεται στην έξελα και αλλού είναι η ενίσχυση του ρόλου των φορέων τοπικής και περιφερειακής αυτοδίκησης στην ε, υλοποίηση των πόρων των ταμείων, ιδίω του Ταμείου Αλία. Και τέλο, τρίτη κατηγορία τροπολογιών που με απασχολεί είναι αυτέ που επιμένουν στην πολιτική βιωσιμότητα ε, των πόρων, των αποθεμάτων δηλαδή και τη διατηρήση της βιοποικιλότητας. Αυτές είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την εκταμείευση και την απόδοση των κοντιλίων. Να εντοπίσω και ένα πρόβλημα ολοκληρώνοντα ε, πολιτικού χαρακτήρα περισσότερο, που το συζητήσαμε και στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Αυτό του άρθρου 3. Με συγχωρείτε, του άρθρου 21. Το οποίο θέτει μακροοικονομικές ε, προϋποθέσεις, την αιρεσιμότητα, επιβάλλοντας την αυστηρή δημοσιονομική πειθαρχία και στις περιφέρειες. Η Επιτροπή προτείνει κυρώσεις για τις περιφέρειες εάν πληρώσουν εντό εισαγωγικών, γιατί τα κράτη-μέλη έχουν κάνει κάποιες, έχουν παραβεί το αυστηρό δημοσιονομικό πλαίσιο. Αυτό δεν μας φαίνεται λογικό και γι' αυτό στην τροπολογία 7 προτείνουμε την άρση αυτής της μακροοικονομικής ερεσιμότητας. Σα ευχαριστώ. Ελπίζω να έρθουν στα χέρια μου γρήγορα τροπολογίες. Εάν είμαι καλά ενωμηρωμένος πρόεδρε, θα μα πείτε κι εσεί πότε λέγεται αυτή η προθεσμία. Ναι, όντω, λίγη στι 4 Ιουνίου η διορία για τι ε, τροπολογίε. 4 Ιουνίου το μεσημέρι. Ευχαριστούμε κύριε Μπεσέ. Το λόγο ζήτησε ο κύριο Καντέ. Καλώς κανεί. Ο κ. Καντέκ. Καταρχήν να ευχαριστήσω τον Ζαν Πολ για την πολύ αξιόλογη γνωμοδότησή του και να υπενθυμίσω ότι στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπου εξετάζουμε το Γενικό Κανονισμό, αντιταχθήκαμε στην μακροοικονομική αιρεσιμότητα. Γιατί θα επιβάλλει διπλή κύρωση ουσιαστικά στις εν λόγω περιοχές το ίδιο θα πρέπει να κάνουμε και στη δική μας γνωμοδότηση, να ταχθούμε κατά της μακροοικονομικής αρεσιμότητας. Είναι λογικό, συνεπές και δίκαιο. Ευχαριστώ. Και τέλος, να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αν θέλει. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον συντάκτη γνωμοδότηση, τον κύριο Μπεσέ, για την μεστή του έκθεση και να πω ότι συνάδει πλήρως με την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί υιοθετεί την ε, ολοκληρωμένη εστίαση, της, ε, το, στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης και την εδαφική ολοκλήρωση. Νομίζω ότι ήταν σημαντική η συμβολή του συντάκτης γνωμοδότησης ως προς την συγκεκριμενοποίηση του ορισμού του στόχου της προστασίας του περιβάλλοντος, ορίζοντας ε, και συμπεριλαμβάνοντας τον ορισμό και την ε, βιοπικιλότητα, εξηγώντας τι θα πει οικονομία με χαμηλή χρήση άνθρακα. Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό το στοιχείο ήδη περιλαμβάνεται, καλύπτεται από την πρόταση. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος όμως κατέθεσε παρόμοιες τροπολογίες Και μια και δεν είναι θέμα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα δούμε πώς θα συνδυαστούν οι διάφορες τροπολογίες από τις ε, αρμόδιες επιτροπές και πώς θα διαμορφωθεί η συζήτηση στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Τώρα η πρόταση για την αντικατάσταση της ανάπτυξης, της εφιούς ανάπτυξης ε, ε, που περιλαμβάνει και δεν αποκλείει και θα είναι και βιώσιμη Ε, η αντικατάσταση αυτού του όρου ε, αφορά περισσότερο φιλοσοφικές ε, θέσεις που όμως δεν είναι άμυρη συνεπειών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίμησε να εφαρμόσει για την μεγέθυνση, την οικονομική ανάπτυξη ως βάση τη στρατηγική ορίζοντας 2020. Προς το παρόν δηλαδή δεν θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τροποποιήσει αυτή τη διατύπωση. Παρόλο που καταλαβαίνουμε γιατί ο εισηγητή προτείνει διαφορετική διατύπωση. Σε ό,τι αφορά τη μακροοικονομική αιρεσιμότητα, σίγουρα αυτό το θέμα είναι νευραλγικό, βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας περίοδου προγραμματισμού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιλαμβάνεται την επιχειρηματολογία και του συντάκτη γνωμοδότης, αλλά και άλλων επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σε τελική ανάλυση πρόκειται για ένα συμπληρωματικό στοιχείο. Προστίθεται στους μηχανισμούς και τις διατάξεις που στόχο έχουν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα της εκτέλεσης και τον αντίκτυπο των δράσεων των ταμείων. Βέβαια, τα πλεονεκτήματα αυτά εμπεριέχουν και κάποιες, ε, κάποια μειονεκτήματα, γιατί καθιστούν υπεύθυνε τις α, ε, τοπικές αρχές. Στη διάρκεια της συζήτηση όμως ε, θα αναλυθούν όλα αυτά τα θέματα πιο διεξοδικά. Βρισκόμαστε στην αρχή των διαπραγματεύσεων. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν αυτές. Πάντως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι στη διάθεση της Επιτροπής σας για περαιτέρω συζητήσεις και διευκρινήσεις. Ευχαριστώ. Θέλει έως κανείς το λόγο. Όχι κανείς. Πολύ ωραία. Οπότε ολοκληρώνουμε τη σημερινή μα συνεδρίαση. Αύριο θα ξεκινήσουμε 9 ακριβώ με τη συνεδρίαση των συντονιστών. Σας ευχαριστώ θερμά, ευχαριστώ και τους διερμηνείς και αύριο με το καλό, αν ο Θεός.